μέχρι τις 11 το βράδυ. Η ατζέντα και το πρόγραμμα έχουν δημοσιευτεί και είναι στη διάθεσή σας και στο δίκτυο, στην σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος της συνεδρίασης.